στην ψηφοφορία. Αντίο κύριε Επίτροπε, τώρα θα υποδεχτούμε την κυρία Γεωργίευα, γιατί θα περάσουμε στην έκθεση Στρίλφερ, Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Πού είστε κυρία Στρίφλερ? Εκεί πάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς ε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργίευα για τη δέσμευση, για τις προσπάθειές της, για τη δημιουργία αυτής της νέας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της Συνήκης της Λισαβόνας ε, και να τονίσω ότι είχαμε πολύ στενή συνεργασία και εξαιρετική συνεννόηση σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Επίτροπε. Στόχος είναι λοιπόν με αυτή την πρόταση να προβάλλουμε τις ανθρωπιστικές αξίες, την αλληλεγγύη της Ένωσης, σε άτομα που είναι σε ε, Δύσκολε συνθήκε, βελτιώνοντα τι δυνατότητε τη Ένωση να ανταποκρίνεται σε ανθρωπιστικέ κρίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει την κατάλληλη ανθρωπιστική βοήθεια εν ώψη της αύξησης ε, ε, του εύρου και του αριθμού των ανθρωπιστικών κρίσεων. Οι εθελοντές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και άλλων, ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ κατεπίγουσα βοήθεια, ανοικοδόμηση, ανάπτυξη. Όλα θα γίνουν για να μπορέσουν οι εθελοντές να προσφέρουν προσφέρουν μια πραγματική προστέμενη αξία. Γιατί θα αναπτύσσονται δυνάμει των ε, αναγκών που θα αναγνωρίζονται επί τόπου και θα έχουν σαφή ρόλο και θα είναι συμπληρωματικοί ουσιαστικά ω προ τι δομέ και οργανισμού που ήδη υπάρχουν και, για την βέβαια και η ασφάλειά του δεν είναι εγγυημένη. Κάθε ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να δηλώσει. Ε, ότι θέλει να είναι θελοντής σε μια τέτοια διαδικασία και οι και συνταξιούχοι και άλλοι πέραν της αξιολόγησης της εμπειρίας αυτών των εθελοντών με επιστοποίηση ε, μετά την ανάπτυξη του επιτόπου θα αποκτούν λοιπόν τις τα απαραίτητα διαπιστευτήρια σε πιλωτικές δράσεις ε, βλέπουμε ότι ε, οι εθελοντές αποκτούν σημαντικές ε, εμπειρίες βοηθώντας ενδεείς ομάδες. Επίσης πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα συμπληρώσει κενά στο τομέα του ανθρωπιστικού εθελοντισμού και θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης και στην ιδέα της ευρωπαϊκή ηθαγένειας. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι επιτακτική ανάγκη ηθικής φύσεως. Λυπούμε βέβαια που ο προπολογισμό για την περίοδο 14-20 μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν και έτσι βέβαια μειώνεται και ο αριθμό των εθελοντών που θα αναπτυχθούν. Και επειδή έχω το λόγο, ε, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου, γιατί η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ δεν έχει απαραίτητα μέσα στη διάθεσή τη για να καλύψει τι αυξανόμενε ανθρωπιστικέ ανάγκε. Γνωρίζουμε τα προβλήματα με την καθυστέρηση πληρωμών για το ΕΚΟ. Είμαι βέβαια ότι η πρωτοβουλία αυτή θα επιτύχει ώστε να βοηθήσει τα πλέον ευάλωτα άτομα. Και γι' αυτό το στόχο, ε, η συμμετοχή ε, των εθελοντών και αυτής της πρωτοβουλίας και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ε, θα είναι σημαντικό στοιχείο και βέβαια όλα αυτά θα τα αξιολογούμε σε τακτά διαστήματα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Στριφλέρ και δίνω το λόγο στον Επίτροπο Γεωργίεβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κυρία Στρίφλερ για την σταθερή και συνεχή στήριξη της για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας. Εδώ πέρα αντικατοπτρίζονται οι επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών, τους οποίους εκπροσωπείται σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, 88% των Ευρωπαίων είναι υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου σώματος και θέλουν να συσταθεί αμέσως με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου. Καταλήγουμε τώρα στην τελική φάση δηλαδή την υλοποίηση της επιθυμίας τους και ως αποτέλεσμα αυτού μέχρι το 2020 γύρω στους 20.000 Ευρωπαίους θα έχουν λάβει μέρος που θα ωφελούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη και όπως είπε η κυρία Στρίφλερ δυστυχώς ο αριθμός τους αυξάνεται αλλά επίσης θα ωφεληθούν και οι ίδιοι οι εθελοντές με το να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εμπειρίες σε αυτή τη φάση των σφιχτών προπολογισμών. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να αξιοποιούμε σωστά τα χρήματα, να συμπληρώνουν οι Ευρωπαίοι θελοντές τα υφιστάμενα σχήματα και να τους βοηθήσουμε και αυτούς. Οι περισσότεροι είναι νέοι και για αυτούς ο εθελοντισμός είναι ένας ε, τρόπος να γίνουν πιο ανταγωνιστική σε μια πιο δύσκολη αγορά εργασίας. Έχουμε τρεις γύρους πιλωτικών έργων ε, με πάνω από 40 ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις για να δούμε το τι χρειάζεται όσον αφορά τις προδιαγραφές στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη για να πετύχει το πρόγραμμα τον στόχο του να είναι δηλαδή μια πλατφόρμα έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να ζήσουν τις αξίες τους, να βοηθήσουν αυτούς που το χρειάζονται. Και είδαμε τον ενθουσιασμό όσων έλαβαν μέρος πάνω από 250 άτομα από νέους μέχρι τους ε, νέους στην καρδιά. Ο νεότερος ήταν 21, ε, ο πιο όριμος ήταν 70. Και ειλικρινά όταν τους συναντάω αισθάνομαι υπερήφανη που είμαι η Ευρωπαία Επιτροπής Ανθρωπιστικής Βοήθειας γιατί ε, αποδεικνύουμε πως δεν είναι τυχαία η Ευρώπη παγκόσμιος ηγέτης αυτό συγκεκριμένα τώρα για τις συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να τονίσω κάποιες από αυτές. Το Κοινοβούλιο έχει θέσει την ενεργό Ευρωπαϊκή Ιθαγενεία ως ένα στόχο της πρωτοβουλίας αυτής. Το Κοινοβούλιο ε, είπε πως θα πρέπει η ασφάλεια των εθελοντών πρώτη προτεραιότητα. Οπότε δεν θα αναπτυχθούν σε θέατρα ενοπλών συγκρούσεων. Ανταυτού δώσαμε βάση σε όσους δουλεύουν σε αντιμετώπιση καταστροφών, ανακούφιση, ανάπτυξη και βεβαίως αυτή είναι το μίσο που υπάρχει και έλλειψη δεξιοτήτων σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Τέλος, το Κοινοβούλιο πρόθεσε τη διάσταση του φύλου σε συνεργασία με γυναίκες. Και όποτε πάω σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές, βλέπω τις γυναίκες, όχι μόνο θύματα, αλλά αλλά να βοηθούν και να σώζουν ζωές. Επίσης να πω πως αναγνωρίζουμε πως είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Και βεβαίως αναμένουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εφαρμογή του προγράμματος, της ε, πράξης κατά εξουσιοδότηση, στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και στην χρηματοδότηση όπως είπε η κυρία Στρίφλερ και στις ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή και την αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πέτροπε. Τώρα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών η κυρία Μουνίση Δορκίσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν έχουμε 6 εκατομμύρια νέων που είναι κάτω των 25 και ένα εκατομμύριο αυτών είναι στην Ισπανία, καταρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων και αυτή η πρωτοβουλία ενό πανευρωπαϊκού μηχανισμού για ευρωπαϊκό σώμα εθελοντών ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι καλό, καθώ θέλει να αναπτύξει τι ικανότητε και την απασχολησιμότητα των νέων στο ανθρωπιστικό τομέα με τα 147,9 εκατομμύρια ευρώ που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό προβλέπεται να καταρτιστούν 20.000 νέοι και νέοι και 7.000 ντόπιοι. Είναι λιγότερα από αυτά που ζητούσαν η Κομισιόν που ζητούσε 210 εκατομμύρια ευρώ. Το είπε η κυρία Στυλίφλερ, η όμως αν αυτά τα κονδύλια μεταφραστούν σε θέσεις εργασίας για τους νέους τα είναι καλοδεχούμενα. όμως εδώ όλοι συμφωνούμε ότι είναι κάτι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Σκοπιά της Επιτροπής Προπολογισμών η χρηματοδότηση του σώματος αυτού δεν θα γίνει εις βάρος ε, των ε, ταμείων ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια, ούτε θα είναι ανταγωνιστικά με τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελόντων Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουλάν για ένα λεπτό για την ε, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν είναι εδώ. Λοιπόν, εφόσον λείπει θα περάσουμε στον κύριο Κασμαρέκ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο και την εισηγήτρια για την εμπλοκή τους ε, σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια είναι μία από τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα ο ρυθμός των ανθρωπιστικών κρίσεων ε, αυξάνεται και πρέπει να αναλάβουμε κατάλληλη δράση. Πολύ συχνά χρειάστηκε βοήθεια ταυτόχρονα σε πάρα πολλούς τόπους. Η όλη έννοια της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, είναι κάτι το υπέροχο. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαν. Όμως, ε, προκειμένου να απαντήσουμε αποτελεσματικά, πρέπει να έχουμε καλό συντονισμό. Εξού και η ιδέα της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελόντων Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ικανότητά μας να αντιδράσουμε σε ανθρωπιστικές καταστροφές ε, είναι πάρα πολύ καλά αναπτυγμένη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους ε, στις περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα συστήματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν μπορούμε να έχουμε επικαλύψεις δομών. Θα πρέπει να δούμε ποιες αρχές πρέπει να ισχύουν, αρχές που θα διέπουν την ανθρωπιστική βοήθεια αυτή καθεαυτή, όπως ε, παραδείγματο χάρη η συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να δημιουργήσουμε προσθέμενη αξία σχετικά. Ευχαριστώ κυρία Κρέτσου για ένα λεπτό εγώ ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ με τη σειρά μου την κυρία Στριφλέρ για την έκθεσή της. Να συγχαρώ ε, και την κυρία Γεωργίευα για την ε, σταθερή υποστήριξή της ε, προς τη σύσταση αυτού του, του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, που είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μεγαλύτερη προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνέ προσκήνιο για την μετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτε χώρε. Οι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα ανταποκρίνονται στην ανάγκη μα να δείξουμε αλληλεγγύη ε, σε ανθρώπου που αντιμετωπίζουν δυσκολίε και είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, ιδίω σε αυτόν τον καιρό που έχουμε αύξηση φυσικών καταστροφών και μεγάλη οικονομική αστάθεια. Κάτι που σημαίνει ότι δαπανώνται πολύ λιγότεροι πόροι για την ανθρωπιστική δράση. Το να έχουμε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε 5.000 περίπου εθελοντέ ε, που θα αναπτυχθούν για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο και ένας καλός τρόπος για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο ε, Νιούτον Ντάν για τρία λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπω και όλοι οι άλλοι, και εγώ είμαι περήφανο που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση, διότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι καινούριο αυτό το οποίο δρομολογείται και ίσως δεν έχει πάρει τόση ε, ε, προβολή από τα μέσα ε, που θα έπρεπε όμως. Προβλέπεται από την συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι μια πολύ θετική και από πολύ καιρό αναμενόμενη νέα πρωτοβουλία ε, στην Επιτροπή μας ένας μόνο ήταν κατά, οι περισσότεροι, η ψηφιτρική πλειοψηφία ήμασταν υπέρ και η συγκεντρεύει κυρία Στριφλέρ. Άκουσα, ε, όπως και η ίδια και άλλα μέλη της Επιτροπής, ε, τους νέους που συμμετείχαν σε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την εμπειρία που αποκόμισαν, γιατί δεν βοήθησαν μόνο ατυχείς ε, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές, ε, σεισμούς, πλημμύρες κτλ, αλλά βοηθούν τον κόσμο να γίνει καλύτερο καλύτερο μέρος και είπαν επίσης ότι ήταν και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία γιατί συνεργάστηκαν με άλλους ανθρώπους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι μια καθόλου θετική εμπειρία και για μένα είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα, όπως και το πρόγραμμα Εράσμους που επιτρέπει σε φοιτητέ να σπουδάζουν σε διαφορετικά μέρη τη Ευρώπη, να γνωρίζουν άλλου νέου, ε, να μαγειρεύουν σπαγκέτι, ροσμπίφ κτλ. Μπορεί να είναι διαφορετική κουζίνα, αλλά μοιάζουμε. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευτυχεί να βρισκόμαστε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Συμμετείχα ε, στον τριμερή διάλογο και στι προσπάθειε επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο. Και κάτι το οποίο με απογοήτευσε και όχι μόνο και του συναδέλφου μου, ήταν ότι από πλευρά Κοινοβουλίου αυτό που θα θέλαμε θα ήταν οι εθελοντές να έχουν ένα είδος ταυτότητας που να δείχνει ότι αυτό είναι ένα σώμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κονκάρδα με ένα τισέρτ. Ε, τα μέλη του Συμβουλίου όμως ε, θεώρησαν ότι είναι κακή ιδέα και θα πρέπει να ντρέπονται αυτά τα μέλη του Συμβουλίου που θεώρησαν ότι αυτό είναι ε, κακή ιδέα. Γιατί θα έπρεπε οι θελοντέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρουν μαζί του την Ευρωπαϊκή σημαία όπου και αν πηγαίνουν. Αυτό που είπε και η κυρία Γεωργίου είναι πολύ σημαντικό. Που λέει το Ευρωβαρόμετρο, δηλαδή το 88% των πολιτών στην Ένωση είναι υπέρ αυτή τη πρωτοβουλία. Και φυσικά και θα έπρεπε και καλωσορίζω αυτό το αποτέλεσμα. Στη χώρα μου με αυτό το τέρας, ε, το κόμμα UKIP ε, που είναι σε όλα αντίθετο ε, κατά της ευρωπιστικής βοήθειας, κατά των μεταναστών, κατά των αλλοδαπών. Φυσικά και δεν είναι εδώ για να συμμετάχουν στις συζήτηση, δεν με εκπλήσει καθόλου αυτό. Αύριο όμως θέλω να δω τι θα κάνει το UKIP και τα άλλα ευρωσκεπτιστικά κόμματα, θα καταψηφίσουν αυτή την πρόταση, γιατί είναι κάτι πολύ ειδικό, κάτι πολύ καινούριο. Και Ίσως είμαστε λίγοι, πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, αλλά είμαστε υπερήφανοι, όπως είπαν και άλλοι πολλοί συνάλφοι, ε, που είμαστε σε αυτήν ε, την απαρχή, στην ε, δρομολόγηση αυτής της πρωτοβουλίας που θα είναι πολύ ευεργετική για την Ευρώπη και για τον κόσμο εν Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Νιούτον Ντάν. 1,5 λεπτό κύριο Βένσον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο και την κυρία Στρίφλερ. Είναι εξαιρετικό το ότι φτάσαμε τόσο μακριά ώστε είμαστε τώρα στα πρόθυρα της λειτουργίας ε, αυτού του σώματος. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας. Κάποιοι θα πούνε, μα δεν πρέπει να μπλέκεται τώρα με αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ διαφωνώ δεν θεωρώ πως ε, κανείς δεν μπορεί να πει πως δεν θα πρέπει να εμπλακούμε. Είναι ένα ζήτημα αλληλεγγύης, ένα μήνυμα του πως ε, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μέλος της διεθνούς κοινότητας. Αυτό είναι μέρος του ήθους μας ε, και κομμάτι της συνθήκης της Λισαβόνας που μας ικανοποιεί. θα υπάρχει ένα κατάλογο ειδικών εκ των προτέρων. Δεν χρειάζεται να ψάχνει κανείς του ειδικού τελευταία στιγμή. Ακούσαμε ήδη πόσο καλά πήγαν τα πράγματα στις Φιλιππίνες. Ένα θετικό παράδειγμα. Και νομίζω πως ε, προχωράμε στο μέτωπο της διεθνούς βοήθειας. Να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια, την Κομισιόν και όλους του συναδέλφους είναι ένα σημαντικό βήμα για την αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κορτας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στρίφλερ αλλά και την Επίτροπο Γεωργίευα για όλη την υποστήριξη της ομάδας μας. Χαίρομαι για αυτό πολύ σημαντικό βήμα που κάνει το Κοινοβούλιο με την ψηφορία αυτού του κανονισμού γιατί είναι ένα γιγάντιο βήμα λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζητάμε από το 2006 και από το 2009 ε, έγινε υποχρεωτικό με τη Λισαβόνα. Τώρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα Εράσμους αλληλεγγύης. Θα δώσουμε τώρα την ευκαιρία σε εκατοντάδες Ευρωπαίους και σε ειδικό προσωπικό και σε οργανώσεις να καταρτιστούν για την παροχή βοήθειας. Θα υπάρχει Επίσης, συμπληρωματικότητα σε σχέση με τη δουλειά που γίνεται επί τόπου. Θα υπάρχει προσθεμένη αξία στο έργο των εθελοντών και θα ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ αρρωγής αποκατάστασης και ανάπτυξη. Αλλά θα έχουμε και άλλα πλεονεκτήματα. Οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να αναλάβουν τις δεσμεύσεις τους ως προς την ελληνική και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θα έχουμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία. Επίσης, ε, θα είναι ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που υπάρχουν περισσότερε ελλείψεις και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πιο αλληλέγγυη Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Κορτές, ο κύριος Πρέντα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Στρίφλερ για την έκθεσή της και να πω ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να πετύχουμε τα όσα δηλώνονται στο άρθρο 214 της Δυτικής της Λαβώνας, δηλαδή να εφαρμόσουμε το πλαίσιο έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ πλήρως με την εισηγήτρια ότι οι δράσεις των μελών του Σώματος Εθελοντών θα πρέπει να βασίζονται στην ανθρωπιστική, στη συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες που έχουν εντοπιστεί τοπικά. Επίσης, αποκλείω και εγώ την περίπτωση παρέμβασης ε, σε ένοπλες σειράξεις. Θα πρέπει να εγγυθούμε την ασφάλεια των εθελοντών. Καλωσορίζω τη συμπερίληψη της ρήτρας αναθεώρησης ε, που έχει συμπεριληφθεί κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου. Αυτό θα μας βελτιώσει, θα επιτρέψει, με συγχωρείτε, να βελτιώσουμε το σύστημα και είμαι πεπισμένο ότι αυτό το νέο νομοθέτημα θα βελτιώσει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοηθείας ε, θα δέσει σε εφαρμογή τις ανθρωπιστικές μας αξίες και αυτό θα δώσει στους νέους την ευκαιρία να δείξουν την αλληλεγγύη τους σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε τρίτες χώρες. Αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Θελοντών φυσικά θα βελτιώσει την ανθρωπιστική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα την κάνει πιο αποτελεσματική. Κύριε Παπαδοπούλου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, European Voluntary Humanitarian Aid Corps has already been... Το το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστική Βοήθεια είχε προταθεί ήδη από την Κομισιόν το 2012 για να εκφράσει τι ευρωπαϊκέ αξίε αλληλεγγύη σε όσου αντιμετωπίζουν ε, ανθρωπιστικές καταστροφές και ανθρωπογενείς ε, κρίσεις. Ε, τώρα λοιπόν σκοπεύουμε να συσταθεί το σώμα αυτό για να συμπληρώσει τις υφιστάμενες δομές και να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη. Έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε, να εκπαιδεύσουμε και να αναπτύξουμε εθελοντές σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και επίσης ε, εισάγεται εδώ πέρα μια αξιολόγηση των εθελοντών αυτών με βάση συγκεκριμένους δείκτες. Προσωπικά είμαι υπέρ των ποσοτικών και ποιοτικών δικτών για τον κάθε επιχειρησιακό στόχο. Συγχαρητήρια για την πρόταση. Μάλιστα, περνάμε στο KTI. 11 ετήματα έχουμε. Θα δώσω λόγο σε όλους. Παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Ένα λεπτάκι και τέλος. Η κυρία Παναγιώτα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την πρόταση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Σώματο Εθελοντών Ανθρωπιστική Βοήθεια. Θέλω να συγχαρώ και την Επίτροπο Γεωργίευα, που είναι συνεπεί στι προσπάθειέ τη ε, για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία αυτή. Κάτι που θα εγγυηθεί και την επιτυχία του σώματο. Θυμάμαι όταν πριν από δύο χρόνια εκπροσώπησα την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου Είχαμε τότε την ε, υποστήριξη των κομμάτων για την δημιουργία αυτού του σώματος εθελοντών και σίγουρα μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων, να τους παράσχει δυνατότητες για να σπουδάσουν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να συμπεριληφθούν στα δίκτυα, στα μητρώα των Ευρωπαίων εθελοντών. Χαιρετίζω την πρόταση για την αναγνώριση του εθελοντικού έργου ως επαγγελματική εμπειρία. Διακόπτεται Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Θεωρώ πως η σύσταση αυτού του σώματος είναι πάρα πολύ σημαντική για, και για τους Ευρωπαίους νέους ε, τους δυνατότητα να πάνε στις χώρες που όπου χρειάζονται να συλλέξουν εμπειρίες και θα δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς να νιώσουν την πραγματική φτώχεια και την πραγματική ανάγκη γιατί στην Ευρώπη υπάρχει μια νοοτροπία των απαιτήσεων δηλαδή όλα τα θεωρούμε αυτονόητα στέγη, τροφή, σχολείο και να βασιζόμαστε στους άλλους όταν αρρωσταίνουμε, είμαστε άνεργοι και γερνάμε. Νομίζω θα είναι και μια επαφή με την πραγματικότητα και θα το κάνει καλό. ευχαριστώ Νικολάζικ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η πρόταση για έναν κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους για όσους έχουν ανάγκη. Είναι θετικό το ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ε, βοηθούν προσωπικά όσους χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει όμως να δούμε και ποιες θα είναι οι συνθήκες τόπου. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ασφαλείας. Εντάξει, καλή καλή καρδιά, αλλά θα πρέπει και ο νομοθέτης να σκύψει πάνω από το ζήτημα. Ευχαριστώ, Φερέρα. Το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν αμφισβητούμε το αντίθετο. Ε, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα συναισθήματα αλτρουισμού και γενοδορίας που έχουν πολλοί Ευρωπαίοι και θέλουν να γίνουν εθελοντές υπό πολλέ διαφορετικές μορφές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως, ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούμε εδώ παρά να μην εκφράσουμε κάποιες επιφυλάξεις για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Εδώ βλέπουμε ότι ε, αυτή η οπτική θέλει να εκφράσει μέσω του θελετισμού κάποιες αξίες και συναισθήματα που δυστυχώς δεν είναι παρόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στις τομέακες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μάλιστα κάποιες από αυτές τις πολιτικές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και γενικά εδώ δεν θεωρούμε ότι συνεισφέρουμε για την ενίσχυση της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Έχουμε κάποιες ανησυχίες λοιπόν του είδους και θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Όπως είπε ο κύριος Νιούτον ε, Ντάν, προλίγου ε, είναι ότι όταν γίνεται κάτι καλό δεν ακούγεται πάρα πολύ στα ΜΜΕ και είπε και ε, η Επίτροπος ότι το 90% των Ευρωπαίων πολιτών είναι υπέρ τέτοιων προτάσεων ε, και νομίζω θα πρέπει να υποστηρίξουμε την εισηγήτρια και τους συναδέλφους τους για την πολύ καλή δουλειά προκειμένου να μας παρουσιάσουν αυτές τις προτάσεις. Φυσικά είναι πολύ καλή ιδέα να θέλουν οι άνθρωποι να εργαστούν εθελοντικά. Ξέρω αρκετούς ανθρώπους που έχουν κάνει θελοντική δουλειά, αφού ολοκληρώσαν τις σπουδές τους και πήγαν στο εξωτερικό για να προσφέρουν τέτοιε υπηρεσίες εθελοντισμού. Επίσης, ε, ξέρω και άλλους ηλικιωμένου ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί και περνούν πολύ από το χρόνο τους εργαζόμενοι ως εθελοντές. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα να οργανώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να μπορούν να εργαστούν μαζί. Ευχαριστώ. Κύριε Σόμπερμαϊρ θα ήθελα να πω το εξή στο συνάδελφο που λέει πως δημιουργούν προβλήματα. Μπορεί να ασκεί κανείς κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να θέλει να βοηθήσει. Μπορούμε να είμαστε θελοντές πυροσβέστες. Εγώ προσωπικά Είμαι, και δεν χρειάζομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχα πάει και στην ε, Ιταλία να βοηθήσω σε πυρκαγιές κτλ. Η πρόταση είναι καλή, ναι, καλό είναι να παρακινήσουμε τους νέους να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να πω και κάτι θετικό να υπενθυμίσω πως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και εντός της Ευρώπης. Έχουμε κράτη-μέλη που δεν κάνουν καθόλου πρόληψη. Π.χ. στην Ελλάδα πρόληψη, προληπτική δράση όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Δεν υπάρχει καμία. Εκεί πέρα μπορούν να πάνε οι νέοι μας. Σας ευχαριστώ κυρία Σουίκα. Σας ευχαριστώ. Όπως είδαμε προσφάτως όταν χτυπάει η καταστροφή χρειάζεται να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί για να βοηθήσουμε τα θύματα με το να βοηθάμε αυτούς τους πληθυσμούς βεβαίως ανταποκρινόμαστε και σε μια ηθική επιταγή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το 50% της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας και εδώ πέρα βεβαίως προβλέπεται η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 85% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν πως είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια ακόμα και σε καιρούς κρίσης. Τη στιγμή που μιλάμε γι' αυτά, στην Κροατία 466 ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, δραστηριοποιήθηκαν το 2012 στο πρόγραμμα αυτό με αρκετούς εθελοντές. Οπότε υπάρχει νομίζω και στην Κροατία αρκετά εκτεταμένος εθελοντισμός crizele umanitare înregistrate în ultimii ani la nivel mondial impun o Οι ανθρωπιστικές κρίσεις απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί εντατικότερα για να βελτιστοποιήσει την αντίδρασή της σε τέτοια φαινόμενα. Η ιδέα του να συστήσουμε ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών ανθρωπιστική βοήθεια είναι συγκεκριμένη έκφραση τη Ευρωπαϊκή Ελληνικής και τη κοινωνική συνοχή στην πράξη. Η ενεργοποίηση των εθελοντών και η κατάρτιση του. Ε, θα προσθέσει αξία στο σύστημα που έχουμε ήδη και η ιδέα ενό πλαισίου για να συνεισφέρουν οι νέοι άνθρωποι σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Θα έχουμε και ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους για τη σημασία του θελοντισμού και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα της συνοχής, ε, της ε, προώθησης, της συμμετοχής στα κοινά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάτουλα. Από την πλευρά των φιλελευθέρων υπάρχει κάποιος συνάδελφος που Μα επισήμανε ότι αφενό ε, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό σώμα εθελοντών και ότι εμεί, ως Ευρωπαίοι θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι υπό τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σημείωσε ότι εμεί, οι ευρωσκεπτικιστέ ε, δεν είμαστε και τόσο της ίδια άποψη. Ελάτε στην Ουγγαρία και θα σα οδηγήσω σε ένα εργοστάσιο σε μια μεγάλη αλυσίδα όπου εργάζονται οι Ουγγροί για 250 ευρώ το μήνα χωρίς κανένα δικαίωμα. Προσπαθήστε λοιπόν να πείστε τους ανθρώπους αυτούς να είναι περήφανοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη σημαία της. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς θα τα καταφέρνατε σε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ κύριο Πλέγκοβιτς. Ένα λεπτό κύριε Μπλεκοβίτ, γιατί υπάρχει μπλε κάρτα. Κύριε Μορβάη δέχεστε. Δέχεστε μια μπλε κάρτα. Ναι. Ευχαριστώ. Κυρία Μορβάη, είναι από την Ουγγαρία η γυναίκα μου και πέρασα στη Βουδαπέστη μέρο από τι διακοπέ των Χριστουγεννιών και έχω οικογένεια στην Ουγγαρία. Έτσι λοιπόν, ευχαρίστω να έρθω στην Ουγγαρία να δεχτώ την προσκλησία σα. Ξέρω πολλού Ούγγρου και ευχαρίστω ε, θα συζητούσα και με πολλού άλλου. Ε, και εγώ νομίζω ότι αυτοί που ξέρω θα ασκούσαν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Κυρία Μορβάη. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ σοβαρή σε ό,τι αφορά την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστώ ε, να ε, σας πάω αν θέλετε να δείτε και τα αξιοθέατα, αλλά απ' την άλλη θα ήθελα να σας πάω ε, και να δείτε και τα εργοστάσια και στο μεγάλο κατάστημα της Τέσκο ή σε άλλα μεγάλα σούπερ μάρκετ όπου οι άνθρωποι εργάζονται για 250 ευρώ και θα ήθελα να πείσετε τους ανθρώπους αυτούς ε, να είναι περήφανοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, σας ευχαριστώ τώρα ο κύριος Πλέγκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας ε, θα είναι μια καλή πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επικροτώ τις προσπάθειες που έγιναν από την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα μέσα σε αυτή την τετραετία. Πιστεύω ότι πλέον ε, υπάρχει αυτό το μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών και η Κομισιόν και με τις διαβλέψεις που είχε με τις ΜΚΟ ακολουθεί αυτά τα βήματα. Χρειαζόμαστε ένα καλό θεσμικό, μάλλον νομικό πλαίσιο, αλλά και δημοσιονομικό πλαίσιο με αυτά τα 150 εκατομμύρια ε, που είπατε ότι έχουμε στη διάθεσή μας, ε, γιατί αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για τις δραστηριότητες για την νεολαία, αλλά και για ε, πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας που έχουν εμπειρία, που έχουν γνώση και θα μπορούσαν και αυτοί να βοηθήσουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δύσκολε καταστάσεις που είναι σε κρίση. Αυτό το σώμα λοιπόν πιστεύω θα δώσει μεγαλύτερη προβολή, μεγαλύτερη δύναμη και θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλη προβολή για την ανθρωπιστική της βοήθεια. Επόμενος ε, ομιλητής, Στίερ. Συμφωνώ με την κυρία Στριφλέρ και είμαι υπέρ αυτή τη ε, πρωτοβουλία ε, για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστική Βοήθεια, που θα επιβεβαιώσει την ηγεσία τη Ένωση στον τομέα τη αναπτυξιακή βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια. 20.000 είναι οι εθελοντέ που είναι καταγεγραμμένοι στην Κροατία και είμαι βέβαιο ότι θα καλωσορίσουν θερμά αυτή την πρωτοβουλία. Όλα αυτά θα συνεισφέρουν και στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής διάστασης για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ταυτότητας, κάτι που χαρακτηρίζεται και από την ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Ε, κάποιοι από εμά πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό όραμα και απ' την άλλη έχουμε τους ε, λαϊκιστές ε, που δεν πιστεύουν και που θέλουν να κλείσουν τα σύνορα για τους ε, νέους με ψηλά προσόντα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά εσείς δεν θέλετε μάλλον να, να βοηθήσετε κάποιους άλλους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά ικανοποιήθηκα πολύ που άκουσα τόσο μεγάλη υποστήριξη να προσφέρεται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Θελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια, δύο σχόλια για να αντιδράσω στις ακουστικά και ένα καταληκτικό σχόλιο. Τώρα για να αντιδράσω στις παρατηρήσεις. Άκουσα κάποιες ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει την ανάπτυξική της δράση και για το αν οι εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε εργαστεί στο να δημιουργήσουμε ένα σώμα εθελοντός όπου οι άνθρωποι θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να βοηθήσουν τους άλλους αλλά για να βοηθήσουν και τους άλλους να βοηθήσουν τον εαυτό τους έχουμε συμπεριλάβει 7.000 και τοπικά εκπαιδευμένους εθελοντές έτσι ώστε να μπορούμε να συνεισφέρουμε και στην ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Δεύτερον, ακούστηκαν κάποια σχόλια σε σχέση με την προβολή και το πώς μπορούμε να γνωστοποιήσουμε στους πολίτες τα καλά νέα. Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά στην πρωτοβουλία αυτή. Μας υποστηρίζει ένθερμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνουμε πιο ορατοί. Αύριο μάλιστα στις 4 ε, το απόγευμα εγώ και η κυρία Στρίβλερ ε, θα έχουμε μια συζήτηση στο Twitter. Αν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε, είστε ευπρόσδεκτοι. Τώρα, για να είμαστε πιο σοβαροί. Είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο να ανακοινώσει κάποιο τα καλά νέα. Είναι πολύ πιο εύκολο ε, να επικεντρώσει την προσοχή των πολιτών στην καταστροφή όταν συμβαίνει και πολύ δύσκολο να γίνει δουλειά για την αποτροπή της. Και αυτό ακριβώ κάνουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια σήμερα αυτό που κάνουμε στην πολιτική προστασία. Δίνουμε και πολύ μεγάλη έμφαση και την επένδυση που κάνουμε στην προετοιμασία, όσο και αν δύσκολο είναι να γίνει, έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα θύματα αύριο. Και ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση με τη σκληρή δουλειά που θα ξεκινήσει από εδώ και πέρα. Γιατί θα πρέπει τώρα να εφαρμόσουμε αυτή την ε, πρωτοβουλία στην στην πράξη. Και θέλω να τονίσω ότι έχουμε πάρα πολύ διευρυμένη υποστήριξη και ε, από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις αρχικά είχαν εκφράσει κάποιο σκεπτικισμό όμως ε, τώρα έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν και έχω την πεποίθηση ότι όσα και να κάνουμε θα βοηθήσουν την Ευρώπη να είναι μία δύναμη του καλού στον κόσμο και εμείς ως Ευρωπαίοι θα προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως ε, μια περιφέρεια που είναι πλούσια όχι μόνο σε πόρους και σε χρήμα αλλά και σε ανθρώπους και σε αξίες. Και αυτό μου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση για τη δουλειά που κάνουμε μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε στρίφλερ έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομη πράγματι. Πρώτα απ' όλα, επειδή τα πάντα έχουν ελεγχθεί θα ήθελα να τονίσω στην αρχή υπήρχαν ορισμένε ε, αμφιβολίες σε σχέση με τις ΜΚΟ σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εθελοντικού σώματος, αλλά από την έκθεση αυτή μπορείτε να διαπιστώσετε ότι έχουμε ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί και έχουμε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Θα ήθελα πράγματι να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες, διότι πρόκειται για μια θαυμάσια προσπάθεια από κοινού εργασίας των σκιωδών εισηγητών. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συνεργάτες μου, την Επίτροπο κυρία Γεώργιεβα, ήταν ένα εγχείρημα το οποίο κράτησε πάρα πολύ καιρό, αλλά νομίζω με τον τρόπο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα νέο εργαλείο, μια προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι αντανακλά πλήρω το πνεύμα τη Ευρωπαϊκής Ιθαγένεια το οποίο χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε κύριε Στρίφλερ. Κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό και αύριο το μεσημέρι θα γίνει η ψήφιση των αρμοδίων ψηφισμάτων. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Στην ημέρα διάταξη έχουμε τώρα τις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Καταρχήν, δίνω το λόγο στον κύριο Νικουλέσκου για ένα λεπτό.